Uh, uh, Καλησπέρα σας λοιπόν. Με χαρά καλωσορίζω στην Επιτροπή μας απόψε και νομίζω μέχρι τις 4.30, αν δεν απατώμε. Τον Επίτροπο για την επιχειρηματικότητα, τον κύριο Ταγιάννη. Έχουμε αρκετά θέματα. από τη Γενική Διεύθυνση για την επιχειρηματικότητα να συζητήσουμε. Σας ενημερώνω, φαντάζομαι ότι σας ικανοποιήσει το ότι ψηφίσαμε σήμερα για την ε, νέα ε, εναρμόνιση των νομοθεσιών. Το πακέτο εναρμόνισης. και επίσης ότι πριν από δύο μήνες υιοθετήθηκε από την Επιτροπή μας ε, το νέο πακέτο για τα πρότυπα που είχε πολύ μεγάλη σημασία πιστεύω ως ε, απόφαση. Περιμένουμε λοιπόν να σας ακούσουμε τι ιδέες έχετε για το μέλλον. Και ειδικά για μια ενιαία αγορά για προϊόντα. Και επίσης εξεργαζόμαστε και άλλες οδηγίες όπως αυτή τη σχετική με τα οχήματα αναψυχής. Αυτά προς το παρόν. Περιμένουμε τις δικές σας ιδέες και προτάσεις. Και ασφαλώς θα υπάρξουν στη συνέχεια και ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Κύριε Σταγιάννη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ξεκινώ. Είχαμε στον Περλεμό μια συνεδρίαση για την χαλιβουργία της Ευρώπης, πολύ σημαντική. Η σημερινή συνάντηση έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα. διότι συμπίπτει, ακολουθεί μετά από λίγες εβδομάδες την έγκριση της νέας στρατηγικής για τη βιομηχανική πολιτική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχα τη χαρά να παρουσιάζω στους σοσιαλιστές και δημοκράτες άλλωστε και στο κόμμα των ε, φιλελευθερών, στο Λαϊκό Κόμμα, συγγνώμη, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την ε, πρόταση αυτή. Έτσι λοιπόν η βιομηχανική πολιτική βρίσκεται πάλι στο κέντρο της οικονομικής μας πολιτικής και της πραγματικής οικονομίας. Και όταν λέμε πραγματική οικονομία προφανώς έχουμε κατά νου και την εσωτερική αγορά. Μια καλή ε, βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική που στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι απαραίτητη ώστε η εσωτερική αγορά να μπορέσει να αναπτυχθεί. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για να καταπολεμήσουμε την κρίση. Ορίσαμε έναν φιλόδοξο στόχο για τα ερχόμενα χρόνια, ώστε μέχρι το 2020 το 20% του εγχώριου εκαθάριστου προϊόντος να προέρχεται από τη βιομηχανική πολιτική. Και αυτό θα είναι δυνατόν εάν γίνει μια σειρά από επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Τομείς προτεραιότητας, ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς, όπως τις ε, τεχνολογίες, τις νανοτεχνολογίες, τη βιοτεχνολογία, τα, τις πράσινες, ε, την πράσινη αυτοκινητοβιομηχανία, τις πρώτες ύλες, τα εφή δίκτυα, Όλα αυτά θα γίνουν εάν δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, γιατί κινητήριος δύναμη της Ευρώπης μπορεί να είναι η μεγάλη εσωτερική της αγορά, με μισό δις καταναλωτών. Καταναλωτές που μπορούν να μας επιτρέψουν να συναγωνιστούμε με την Ινδία και την Κίνα, αλλά εφόσον επενδύσουμε στην ποιότητα της παραγωγής μας. η δική μας ε, δουλειά, η προσπάθειά μας για επιχειρηματική και βιομηχανική πολιτική που να είναι ισχυρότερες βασίζονται σε όσα γίνονται για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Μάλιστα σε συνεργασία με τον Επίτροπο Μπαρνιέ για την υλοποίηση και την εφαρμογή της πράξης για την ενιαία αγορά 1 και 2 των Single Market Act. Και όταν μιλάμε για μηχανική πολιτική, μας ενδιαφέρει προφανώς και η πρόσβαση των επιχειρήσεων στις πιστώσεις όπως τον τομέα του κεφαλαίου κινδύνου, του venture capital ή την υλοποίηση της Βασιλείας 3 ή την υλοποίηση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Η πρόσβαση στις αγορές είναι εργαλείο καθοριστικό για την ανάπτυξη και όταν μιλάμε για την αγορά, εννοούμε κυρίω την εσωτερική αγορά. Υπάρχουν βεβαίω και οι εξωευρωπαϊκέ αγορέ. Και βεβαίω ο κύριο Μόντι, πριν γίνει πρωθυπουργό στην Ιταλία, είχε τονίσει στην σχετική έκθεσή του τα θέματα αυτά. Ποιοι είναι οι φραγμοί που δυσκολεύουν την ανάπτυξη της ε, οικονομίας μας μέσω της εσωτερικής αγοράς. Ένα από τα βασικότερα λοιπόν εργαλεία που διαθέτουμε για την βιομηχανική μας πολιτική και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ευθύ αμέσω τα μέλη της Επιτροπής σας ε, και τους εισηγητές είναι οι νέοι κανόνες για την τυποποίηση. Πριν λίγες εβδομάδες το Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τα ενέκριναν είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να τονίσουμε την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού μας και επιχειρησιακού συστήματος προκειμένου να ερευνήσουμε και να διερευνήσουμε νέες αγορές και να επιβάλλουμε τα πρότυπά μας. Έτσι θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να είναι ανταγωνιστικότερες. Σε περιοχές του κόσμου σημαντικές όπως η Ρωσία, η Λατινική Αμερική, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την τυποποίηση, πρόγραμμα που θα εγκριθεί στο πρώτο εξάμενο το 2013, είναι ένα νέο εργαλείο για να σχεδιάσουμε την δράση σε σχέση με την τυποποίηση και πάντοτε βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει με συγκεκριμένες εντολές να υλοποιηθούν αυτά τα πρότυπα από τους ε, επίσημους φορείς τυποποίησης της Ευρώπης. Υπάρχουν τομεί προτεραιότητα για την τυποποίηση, όπω έχουν εντοπιστεί στην ανακοίνωση για την νέα βιομηχανική πολιτική, προκειμένου να αναπτυχθούν οι υποδομέ και η ψηφιακή αγορά. Τέλο, το ετήσιο πρόγραμμα εργασία τη Ένωση θα συμπεριλαμβάνει και στόχου για τη διεθνή διάσταση, όπω έλεγα προηγουμένω, τη ευρωπαϊκή τυποποίηση. Έτσι θα στηριχθεί η νομοθεσία που επιτρέπει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών πολιτικών. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα τυποποίηση έχουν συζητηθεί πολύ τελευταία. Έχει να κάνει αυτό και με, τα, με την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών, όπως την ε, ηλεκτροδότηση των ηλεκτρικών οχημάτων, την επαναφόρτιση δηλαδή. Αυτό είναι σημαντικό σε επίπεδο διεθνούς αγοράς. Εδώ συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να υπάρξει απαραίτητη πλατφόρμα ή διαπαθή σε ευρωπαϊκό επίπεδο Ήδη πριν από δύο χρόνια ανέθεσα συγκεκριμένη εντολή στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό SENSEN-ELEC για να υπάρξει ένα ενιαίο πρότυπο για, τις, ε, για τους φορτιστές των ηλεκτρικών οχημάτων. Εδώ αναζητήθηκαν συγκεκριμένες λύσεις, αλλά εφόσον εξέπνευσε η εντολή, δεν ε, προέκυψε συμφωνία μέχρι την ημερομηνία λήξης, εκπνοής της εντολής. Έτσι ανέλαβα εγώ ίδιο δράση και ζήτησα από τις υπηρεσίες της Γενικής διεύθυνση να διεξαγάγουν μελέτη αντικτύπου, ώστε να προχωρήσουμε σε νομοθετική πρόταση στις αρχές του επόμενου χρόνου. Δεύτερο παράδειγμα των ενιών φορτιστών. Ακολουθήσαμε το μνημόνιο κατανόησης για το θέμα αυτό και τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει είναι πολύ θετικά βάσει της τελευταίας έκθεσης που έφτασε στα χέρια μας σήμερα, μπορούμε σε έναν κοινό φορτιστή να συνδέσουμε το 90% των νέων μοντέλων ε, ψηφιακών τηλεφώνων που πολλούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό θα είναι, ήταν ήδη εφικτό στο πρώτο εξάμεινο της φετινής χρονιάς. Οπότε η προσπάθειά μας και απέδωσε και ήταν χρήσιμο στους ε, πολίτες της Επίσης, μελετούμε διαφορετικές δυνατότητες η παροχή αυτή, ε, αυτών των υπηρεσιών να συνεχιστούν και μετά την ε, φετινή χρονιά και η συμφωνία να καλύπτει και άλλα ηλεκτρονικά μηχανήματα όπως τα iPad, τους, ε, τα μηχανήματα MP3, τις ηλεκτρονικές κάμερες και ούτω καθεξής. Τώρα, η παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς η πολιτική μας κατεύθυνση ακολουθεί μια βασική αρχή. Ότι πρώτα πρέπει να... Πρώτος ο οποίος θα υποφελείται από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να είναι ο ίδιος ο πολίτης. Έτσι λοιπόν θέλουμε μια ενισχυμένη εσωτερική αγορά στην Ευρώπη, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο της ελεύθερης κυκλοφορίας, α, αλλά και ένα μέσο για να τονωθεί η εμπιστοσύνη που πολλούνται εντός της ευρωπαϊκής ε, αγοράς. Μια ελεύθερη αγορά που κυκλοφορούν ελεύθερα τα αγαθά και τα εμπορεύματα που έχει να κάνει με την παρακολούθηση επίση τη ε, εσωτερική αγορά και του μηχανισμού που χρησιμοποιούνται. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία. Πρέπει να υπάρχει συντονισμό μεταξύ των κρατών, δυνατότητα έγκαιρη παρέμβαση σε όλη την επικράτεια τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ λοιπόν θέλουμε να προτείνουμε μια δέσμη μέτρων που να αφορούν την παρακολούθηση τη αγορά για την ερχόμενη χρονιά. Πρόκειται για μία από τις δράσεις προτεραιότητας που θα προκέπτουν και από την ανακοίνωση για την εσωτερική αγορά, από την, ενία, Brexit για την ενία αγορά νούμερο 2 και την ανακοίνωση για την νέα μηχανική πολιτική. Θα διατηρήσουμε αυτά τα θέματα ως προτεραιότητα. Στη δέσμη αυτή θα περιλαμβάνεται μια πρόταση κανονισμού για την ε, παρακολούθηση της αγοράς, την αναθεώρηση της οδηγίας για την γενική ασφάλεια των ε, αγαθών και ένα πολιετές πρόγραμμα παρακολούθησης ακριβώς. μιας και μίλησα για τα ωφέλη προς τους καταναλωτέ να σταθώ και σε άλλες δύο προτάσεις, ιδιαίτερα σημαντικές και εύστοχε, που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, η... η καταγραφή των οχημάτων σε άλλο κράτος μέλος, πράγμα που αποτελεί ζήτημα κυρίως για τα ηλεκτρικά οχήματα. Κάτι που πολλές φορές ε, παραφέρει, επισύρει μάλλον μεγάλο κόστος. Εδώ έχουμε εντοπίσει τα 20 βασικά πρακτικά προβλήματα των ε, πολιτών σε σχέση με την εσωτερική αγορά. Η κατάσταση δεν μπορούσε να παραμείνει απαράλλακτη γι' αυτό. Και επειδή επιδιώκουμε μια Ευρώπη πιο φιλική προς τους ε, ίδιους τους πολίτες, εντοπίσαμε συγκεκριμένα πρακτικά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση κανονισμού ήδη πριν από κάποιου μήνε, τι αρχέ Απριλίου συγκεκριμένα τη φετινή χρονιά, με στόχο να απλουστευθούν με τρόπο ριζοσπαστικό όλες οι διαδικασίες ε, καταγραφής των οχημάτων σε ένα άλλο κράτος μέλος. Όταν πρέπει η διαδικασία αυτή να επαναληφθεί και αυτό γίνεται με βάση την βασική έδρα, την έδρα κατοικίας ενός πολίτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, που θα μπορεί να επαναληφθεί με μια απλουστευμένη διαδικασία και σε άλλο κράτο μέλος εφόσον υπάρχει ανάγκη. Στις περισσότερες περιπτώσεις η, η τεχνική έλεγχη των οχημάτων θα αντικατασταθούν από την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών για τα διάφορα ηλεκτρικά οχήματα. Έτσι θα αποφύγουν το επιπλέον άχθος οι πολίτες και θα κερδίσουν και χρόνο. Η συγκεκριμένη πρόταση για τους ε, πραγματικούς ελέγχους στα οχήματα θα επιτρέπει και την ε, άρνηση καταγραφής οχήματος. Οπότε θα γίνονται όλα σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την πρόταση το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορούν να μετατρέψουν τις ε, διατάξεις εφόσον χρειάζεται και θα επιτρέψουμε να υπάρξει οικονόμηση μισού δις ευρώ ετησίως. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο και ιδιαίτερα ευαίσθητο για το οποίο θα ήθελα τη στήριξη του Κοινοβουλίου μου είναι και προσφυλές και το θεωρώ και ευαίσθητο θέμα. Γιατί όπως θα θυμάστε από την ακρόαση που είχε οργανωθεί υπήρχε η δέσμευση να τροποποιηθεί η οδηγία αυτή. Η οδηγία για την οδηγία των φαρμακευτικών προϊόντων. Υπήρχε συγκεκριμένο αίτημα της ε, συναδέλφου τη κυρία Γκροστέτ και γι' αυτό υποβλήθηκε πρόταση, νέα πρόταση, στις αρχές Μαρτίου τη φετινή χρονιά. Τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Παρβάνοβα και τον κύριο Μπουζόη για τα σχέδια έκθεσης που στήριζαν ουσιαστικά την πρόταση οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτίθεμε να εργαστώ σκληρά για το θέμα αυτό και, να, και εδώ να τονίσω την ε, επιθυμία μας πραγματικά να ενισχύσουμε τις αρμοδιότητες των κρατών σε θέματα υγείας. Θέλουμε να προλιάνουμε το έδαφος για να καλυφθούν οι ανησυχίες τις οποίες άκουσα με προσοχή το προηγούμενο διάστημα και στο επίπεδο του Κορεπέρ αλλά το επαναλαμβάνω, δεν έχω την πρόθεση, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, να μεταβάλω τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Απλώς θέλουμε να βελτιώσουμε τους ισχύοντες διαδικαστικούς κανόνες. Και εφόσον μιλάμε για ωφέλη για του ε, πολίτε σε σχέση με όλε τι προτάσει περί εσωτερική αγορά που αυτή τη στιγμή συζητώνται, θέλω να επικεντρωθώ και στο εξή. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα πρέπει να μπορούν να υποφεληθούν πλήρω από την ενιαία αγορά. σε τη νομοθεσίας για βιομηχανικά προϊόντα, ένα πρώτο ζήτημα. Η παγκοσμιοποίηση και η καινοτομία έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και στην διοργάνωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών σε πολλές περιπτώσεις. Προϊόντα που πολλές φορές ενσωματώνουν και τεχνολογικά στοιχεία. Οπότε, θα πρέπει να διερωτηθούμε το εξή. Εφόσον είμαστε πεπισμένοι ότι οι κανόνες μας από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα θα μπορούν, να αντιμετωπίσουν ε, τις σημερινές ανάγκες. Ξέρουμε ότι οι σοβαρές εξελίξεις και θα, θα μπορούν να μας διατηρήσουν στην εμπροστοφυλακή των, εξε, ε, νέων καταστάσεων και των μελλοντικών. Εγώ απαντάω όχι, διότι θα μπορέπει να φροντίσουμε να καλύπτουμε τις νέες ανάγκες που προκύπτουν, προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία και βεβαίως εμείς να επικαιροποιούμε διαρκώς και να προσαρμόζουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις τοποθετήσεις των ενδιαφερομένων εδώ, την βιομηχανία, τους καταναλωτές, τις οργανώσεις καταναλωτών επίσης, ε, όσου ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να υπάρχει μια ευρεία σφαιρική προσπάθεια που θα ξεκινήσει ήδη τις ερχόμενες εβδομάδες. Στην αρχή τη παρουσιασή μου μίλησα για το πόσο η εσωτερική αγορά είναι καθοριστικό εργαλείο για, την... για το σχεδιασμό μια βιομηχανική πολιτική που να στηρίζει και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Κατά την άποψή μου είναι ακόμα πολύ φραγμή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπάρχει μελέτη που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τέσσερις εβδομάδες. Αυτό βεβαιώνει ότι το, το γραφειοκρατικό άχθος και η νομική φραγμή ε, αποτελούν τροχοπέδι. Τροχοπέδι που μας ε, ανησυχεί. Δυσκολεύουν την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρεμποδίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες της εσωτερικής αγοράς. Όπως ορίζει και το Small Business Act και αναγνωρίζει και η έκθεση Stoiber για την απλούστευση, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όπως διαρθρώνεται και σε εθνικό επίπεδο, επέτρεψε την εξοικονόμηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και τον περιορισμό του κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως απομένει πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλύψουμε. Ξέρετε ότι σε λίγες εβδομάδες προβλέπεται μια μεγάλη εκδήλωση στην Κύπρο που θα ασχολείται ακριβώς με την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οπότε θα συζητήσουμε και το πώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο την εσωτερική αγορά τα ερχόμενα χρόνια. Δεν μπορούμε παρά να θυμίσουμε ότι είναι σημαντική για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η ανάπτυξη ακριβώς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκατομμύρια τέτοιε επιχειρήσει έχουμε στο έδαφο τη Ένωση που δυσκολεύονται από γραφειοκρατικού φραγμού που θα πρέπει οπωσδήποτε να περιοριστούν. Ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον τομέα τη οδική ασφάλεια. Την 1η Νοεμβρίου τέθηκε σε ισχύ ένας κανονισμός που συνδυάζει 50 παλιές οδηγίες και αφορά την παρακολούθηση της αγοράς και των προϊόντων μεταξύ άλλων. Οι προτάσεις που θα προκύψουν λοιπόν μέσα στην επόμενη χρονιά είναι προτάσεις που θα προβλέπουν και την δύσκολη ερμηνεία με την περίπλοκη αυτή διάρθρωση τόσων οδηγιών που ισχύουν ταυτόχρονα. για να κατανοήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο ποια είναι τα εμπόδια και οι φραγμοί που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, θα διοργανώσουμε γύρω διαβουλεύσεων που θα ολοκληρωθεί περίπου στις 21 Δεκεμβρίου. Σκοπός μας ήταν να εντοπίσουμε εδώ τα 10 βασικά ευρωπαϊκά νομοθετήματα που θεωρούνται εχθρικά προ τη λειτουργία των επιχειρήσεων και εμποδίζουν την ανάπτυξή του. Στο τέλο του γύρου διαβουλεύσεων θα ορίσουμε διορθωτικά μέτρα και προτάσει προκειμένου να καλύψουμε τι ανάγκε των επιχειρηματιών, πάντοτε σεβόμενοι τα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κατά πρώτον, την προστασία των εργαζομένων. Όμως η υπέρμετρη γραφειοκρατία σε κάποιους τομείς κλειδιά πρέπει να περιοριστεί, όπως την παροχή υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο, τις τελενιακές διατυπώσεις, την κατηγοριοποίηση των εμπορευμάτων και του τελενιακούς δασμούς. Στην, ε, στο συντονισμό και την μεταφορά των κοινωνικών δικαιωμάτων επίσης και ένα ακόμη άριστο παράδειγμα για την ε, απλούστευση της νομοθεσίας, η ενέργεια. Εδώ θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη μεγαλύτερη αποδοτικότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα. Μίλησα για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά γνωρίζουμε ότι και τα κράτη-μέλη επιβάλλουν πολλούς κανόνες που και αυτοί δυσκολεύουν κάποιες φορές την ε, εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών συναλλαγών. Όπως ας πούμε την πώληση προϊόντων ενός κάτους μέλους, επιχείρηση ενός κάτους μέλους σε άλλα. Εδώ έχουμε εργαλεία που θα βελτιώσουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και θα επιτρέψουν τέτοιοι φραγμοί να αντιμετωπίζονται εγκαίρως. Να μην παρεμποδίζονται η ελεύθερη κυκλοφορία. Η οδηγία 9834 ακριβώς ε, επιβάλλει στα κράτη-μέλη να κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, όλα, τα άλλα κράτη-μέλη όλα τα προγράμματα και τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ε, προτού ενσωματωθούν στην ε, εσωτερική νομοθεσία. Σκεφτείτε απλώς ότι μόνον πέρσι και φέτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 700 έω 800 εθνικές κοινοποιήσει. Οι δράσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δώσει λοιπόν συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αυτή την περίπτωση. Και όχι μόνο. Στο 95% των περιπτώσεων τα κράτη-μέλη τροποποίησαν τα προγράμματά τους προκειμένου να καλύψουν τις ευρωπαϊκές απαιτήσει και να μην έχουν, ε, να, να έρθουν αντιμέτωπα με διαδικασία παραβάση που και χρονοβόρε είναι και τα πανηρές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες φορές γίνεται λιγάκι χωροφύλακα σε τέτοιε καταστάσεις, όμως νομίζω ότι είναι καλύτερο να υπάρχει διάλογο ε, και θα πρέπει να είναι ίστατη λύση η διαδικασία επί παραβάση, όταν δεν μπορεί να υπάρξει διάλογο και λύση μέσω τη συζήτηση. Έτσι, φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σαν ένα πρόσωπο μηχάνημα που επιβάλλει κυρώσει στα κρατημέλη, μελη Όμω πρέπει να διασφαλίσουμε την καλύτερη διαβίωση των καταναλωτών. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με την εσωτερική αγορά και την εύρυθμη λειτουργία τη. Τον περσινό Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε και έκθεση για το πώ υλοποιείται από τα άλλα θεσμικά όργανα η οδηγία αυτή. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε στα τέλη του χρόνου. Επίσης για την οδηγία 9834 προβλέπουμε και την βελτίωση λειτουργίας της Τράπεζας Δεδομένων Κρίς για να μπορέσουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποφεληθούν καλύτερα από συγκεκριμένες δράσεις. Αυξάνεται συνεχώς και η πρόσβαση, η επιγραμμική πρόσβαση με 300.000 ε, προσπάθειες και κινήσεις έρευνας, μόνο για το 2011 στην Τράπεζα 3. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες μας για τους προσεχείς μήνες προκειμένου να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. Ε, προφανώς δεν έχουμε ούτε καν το χρόνο για να ε, βελτιώσουμε, για να καλύψουμε μάλλον όλες αυτές τις πολυάριθμες ανάγκες που υπάρχουν, αλλά ελπίζω ότι μέσω των ε, ερωτήσεων που θα κάνετε με τη συζήτηση που θα έχουμε εδώ, θα μπορέσουμε να έχουμε μια επικοδομητική και παραγωγική ε, συνεργασία, ώστε να διευκολύνουμε και να κάνουμε λιγότερο γραφειοκρατική την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την διαβίωση των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Well, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε που μοιραστήκατε μαζί μας ένα ευρύτατο φάσμα προτάσεων. Κάποιες δεν τις είχαμε ξανακούσει, κάποιες τις επεξεργαζόμαστε ήδη, αλλά σίγουρα φαίνεται πόσο πολλή δουλειά κάνουμε από κοινού. Για να δούμε λοιπόν πώς προχωρούμε, ποιοι είναι μέχρι στιγμή στον κατάλογο μιλητών, με τη σειρά που ε, σήκωσαν τα χέρια τους. Mr. Salvini, Mr. Arias, Mr. Correa de Campos, Mr. Schaldemose, Mr. Schwab, Mr. Baldessari and Mr. Obermeyer. Now, does anyone miss... Και κυρία Ρουλέ και κυρία Βάιλερ. Tomorrow morning at 10 o'clock meeting. um, European anybody Commission. else who's not on? Okay. Well... Υπάρχει κανένας άλλος? Όχι. Λοιπόν, θα σας κάνω την εξής πρόταση. Θα σας παρακαλέσω να κάνετε ένα σχόλιο του ενός λεπτού και μία σύντομη ερώτηση και θα δίνω το λόγο σε τρεις κάθε φορά και θα φροντίσω και επίτροπος να μην μακρηγόρει στις απαντήσεις του. Κυρία Βάιλερ πρέπει να φύγει, οπότε να την ανεβάσω στον κατάλογο. Διαφωνεί κανείς. Λοιπόν, άρα, πρώτη ομιλητές Κοράτσα Μπίλτ, Χατζημαρκάκης, Βάιλερ. Όχι μαζί με την κυρία Στάιλερ για να μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, κοράτσα μπιλτ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι, Είναι δύσκολο να κάνει σύντομο όμω ε, μετά από αυτέ τι πολλέ ε, προτάσει που ακούσαμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή ε, που δεσμεύτηκε για την απλούστευση, την εναρμόνιση και τη μείωση του άχθου για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Κάτι πολύ σημαντικό σε σχέση με όσα κάνουμε και για τη δέσμευσή σα επίση, κύριε Επίτροπε, σε σχέση με την οδηγία τη καθυστερούμενη πληρωμέ. Ελπίζω λοιπόν να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα του χρόνου. Θέλω να σα κάνω μια ερώτηση για τι εμπορικέ σχέσει μεταξύ επιχειρήσεων Είστε ο πρόεδρος ε, του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την συσφορά στην ε, αλυσίδα τροφίμων και Ξέρετε ότι εγκρίναμε το διάλογο ε, τον πολυτομεακό και το πολυκλαδικό για να έχουμε λύσεις που θα οδηγήσουν σε πιο δίκαιες πρακτικές σε ό,τι αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού σε τρόφιμα. Ιδίω δε θέλουμε να έχουμε μια πιο δίκαιη, ένα πιο δίκαιο λιανεμπόριο βάσει και τη εκθεσή μου. Θέλουμε να έχουμε τα αποτελέσματα μέχρι τα τέλη του έτου. Ακολουθήσατε, βλέπω, και την συνετική λύση, άρα αφήσατε ανοιχτέ όλε τι επιλογέ. Πρέπει να σα πω ότι εμά δεν μα ικανοποίησε το γεγονό ότι ο Επίτροπο ε, Τσόλο ε, μα υποσχέθηκε νομοθεσία, σπάζοντα όμω τη γραμμή που είχατε οθετήσει εσεί και ο Επίτροπο ε, Μπαρνιέ, στηρίζοντα το Κοινοβούλιο. Αλλά τέλο πάντων, αυτό που είναι τώρα σημαντικό είναι και η ανακοίνωση B2B, business to business, που ζητάει το Κοινοβούλιο, και το σχέδιο δράση ε, για το που επίση ζητάει το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε για αυτέ τι διπηρεσιακέ διαβουλεύσει. Μέχρι τα τέλη του χρόνου μα υποσχεθήκατε, ελπίζω, αν και δεν είναι δική σα αρμοδιότητα, ελπίζω να επιταχυνθεί αυτή η διπηρεσιακή διαβούλευση, γιατί θα ήταν πάρα πολύ περίεργο να βάζουμε ένα χρονοδιάγραμμα ε, και διορίες ε, για τους εμπλεκομένους φορείς και μετά να καθυστερεί την παρουσίαση ε, της πρότασης για τι εμπορικέ σχέσει business to business η ίδια η Επιτροπή. Έχουμε το φόρουμ Σύλλογου Εκπαίδευση στι 5 Δεκεμβρίου. Άμα παρουσιάσετε μετά τι προτάσει σα, τότε δεν θα έχουμε εμεί τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Άρα, ερώτημα. Πώ βλέπετε τώρα τη διαδικασία, πώ βλέπετε το μέλλον του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου που λύγει εντολή του στι 5 Δεκεμβρίου. Μπορούμε ίσω με κάποιο τρόπο να εξασφαλίσουμε του εμπλεκομένου φορεί ότι θα υπάρχει μια πιο ανεξάρτητη εποπτεία από του ε, ευρωπαϊκού ε, θεσμού. Πολύ γρήγορα, Ελπίζω να εκτιμήσατε το ότι μίλησα πολύ σύντομα για ένα τόσο πολύπλοκο ζήτημα. Εντάξει, είμαστε πιο έτσι, ανεκτικοί μαζί σας γιατί είστε επικεφαλής για αυτά τα θέματα. Και θα συναντηθώ και εγώ το βράδυ με την κοινοπραξίλια εμπορίου της Βρετανίας, ο κ. Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ, Επίτροπε, κύριε... Ε, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Έχουμε 40 χρόνια ιστορική αγορά, έχουμε τελωνιακή ένωση και διαπιστώνουμε ότι έχει σημειώσει αυτή την εποχή η βιομηχανική παραγωγή πολύ σημαντική μετατόπιση σε περιοχές έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αλλιώς εκεί που δεν υπήρχε μεγάλη παραγωγή εξαφανίζεται ουσιαστικά. Κράτη τα οποία έχουν ε, τη μεγαλύτερη ανεργία, η Ελλάδα και η Ισπανία, ε, είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν το φαινόμενο αυτό πολύ πιο έντονο. Έτσι λοιπόν πρέπει η πολιτική που θα διαμορφώνουμε να έχει μια συνέπεια και συνοχή και γι' αυτό ερωτώ για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε πρόσβαση στη χρηματοδότηση μαζί με τον Επίτροπο Χάν, τον Επίτροπο Ρεν γιατί το σχόλιο μου είναι ότι η χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ μικρή. Έχουμε τρία χρόνια τώρα κρίση με μηδενική δυνατότητα πρόσβαση σε κονδύλια σε χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 11 δις ευρώ που θα μπορούσε ο κύριος Χάν να διαθέσει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για αναπτυξιακά μέτρα, για μέσω αναπτυξιακών τραπεζών κτλ. που δεν κινούνται, δεν διατίθενται, δεν υπάρχει καμία κινητικότητα ούτε στην Ισπανία ούτε στην Ελλάδα. Αυτό είναι η δουλειά μας. Είναι πολύ αρνητικό το αποτέλεσμα. Και ρωτώ λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε για να ξεφύγουμε από την κατάσταση αυτή και να διαθέσετε, να δώσετε μια όθηση στα μέσα αυτά να μπουν στην αγορά. Παραγωγή σε χώρες οι οποίες, σε παραδείγματα, θα μπορούσαν να έχουν φωτοβολταϊκή ενέργεια, δεν έχει γίνει τίποτα. Και για τον τουρισμό. Το quick win δεν θα μπορούσαμε να το στοχεύσουμε με συγκεκριμένα μέτρα για τον τουρισμό. Πρόταση Φερρυπίν 1000 ε, ευρώ πρημοδότηση για κάθε Γερμανό τουρίστα ο οποίος πάει να επισκεφτεί ε, την Ελλάδα ή την Ισπανία. Γιατί όχι. Τρεις ερωτήσεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Δοκιμάσα ε, την υπομονή μου, λέει ο πρόεδρος, η κυρία Βάιλερ. Θα έλεγα για τον κύριο Χατσιμαρκάκη ότι ήταν κατά της πρημοδότησης για την ε, κατάργηση, για την διάλυση των σκαφών. Α, όχι εσείς, ε, γενικά οι φιλελεύθεροι πάντως. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Ταγιάννη, πώς θα έχουν πρόσβαση στην ε, ενίσχυση για τις επενδύσεις, για την ε, ρευστότητα, πώς οι μεγάλες τράπεζες συμπεριφέρονται στην Ευρώπη, γιατί βλέπουμε ότι δεν διαθέτουν ε, κονδύλια, δεν προσφέρουν χρηματοδότηση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και θέλω να ρωτήσω γιατί η ενίσχυση από το Ταμείο Διάσωσης δεν πηγαίνει εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνει. Και επίσης υπάρχει μια ανάλυση για τον λόγο για τον οποίο τα κράτη-μέλη δεν προχωρούν στην ε, ε, εφαρμογή της οδηγίας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Γιατί δεν γίνεται λοιπόν. Όλα τα κράτη είχαν πει το ναι όταν έγινε η πραγματεύση. Ολόκληρο το κοινοβούλιο από την αριστερά μέχρι τη δεξιά πτέρυγα είχαν πει το ναι και τώρα μόνο η Μάλτα και η Κύπρος από ό,τι γνωρίζω έχουν εισαγάγει τη σχετική νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο. Γιατί λοιπόν εδώ πρόκειται για μια ε, για έναν ακρογωνιαίο λίθο της, ε, της ρευστότητας των αγορών μας, γιατί δεν προωθείτε τα μέτρα αυτά, γιατί δεν ελέγχετε την εφαρμογή τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Επίτροπος. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα. Πρέπει να πω ότι πριν πέντε μέρες η Ιταλία μετέφερε την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Τώρα μένουν τρεις χώρες που δεν έχουν υλοποιήσει την οδηγία. Η καταληκτική ημερομηνία, το όριο, είναι ο Μάρτιος του 2013. Ξεκινήσαμε ενημερωτική εκστρατεία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να καταλάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι επιχειρηματίες και οι δικαστές που μετά θα πρέπει να αποφασίσουν για τις κυρώσεις σε περίπτωση που δεν γίνεται σεβαστή οδηγία, προσπαθήσαμε να τους εξηγήσουμε τις λεπτομέρειες της λειτουργίας της νέας αυτής, του νέου αυτού νομοθετήματος. Και σας επιβεβαιώνω ότι ήδη υπάρχουν σοβαρές αντιδράσεις. Ούτε στη χώρα μου δεν ήταν εύκολο να περάσει το μήνυμα, αλλά αυτή τη στιγμή τα ε, κράτη-μέλη πρέπει να πληρώσουν ε, πολλά δις ε, ευρώ στις επιχειρήσεις λόγω των καθυστερήσεων. Δεν είναι απλό λοιπόν να γίνει αποδεκτό αυτό το μέτρο. Βεβαίω νομίζουμε ότι τα οφειλόμενα αυτά χρέη θα πρέπει να αφαιρεθούν από το Σύμφωνο σταθερότητα, Διότι σε πολλά κράτη-μέλη υπολογίζονται στο χρέος αυτές οι οφειλέ, οι εφειλέ του δημοσίου, μόνον όμως εφόσον καταβληθεί η πρώτη πληρωμή. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αρχίσει η καταβολή, δεν περιλαμβάνονται και ως χρέη. Γι' αυτό ζητήσα και από τον ε, αρμόδιο επιτροπό να προβλέψει περιθώριο μετατροπής και, και προσαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας, ιδίως με αυτά που προκύπτουν λόγω των οφειλών προς το δημόσιο από το δημόσιο μάλλον προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόσβαση στις πιστώσεις. Αυτή που ελπίζουμε να υπάρξει, όχι μόνο την ε, ισχύουσα, Ελπίζουμε ότι το σχετικό πλαίσιο θα αρχίσει να λειτουργεί πολύ σύντομα, ήδη από το χρόνο. Ήδη οδηγία για τις καθυστερήσεις περιπλωμών είναι ένα σοβαρό μήνυμα καλεί και τις, τραπεζι, τράπεζες να δίνουν πιο εύκολα δάνεια. Επίσης, ζήτησα τη στηρίξη του Κοινοβουλίου εδώ για, το, για τη Βασιλεία 3 ώστε να μην γίνει ένας καταπιστικός κανόνας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει και ένα φόρουμ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου συμμετέχει και το Ευρωκοινοβούλιο με τους εκπροσώπους του. Και εκεί συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γιατί ούτως ή άλλως οι βιομηχανικές μας πολιτικές σκοπό έχουν ε, να χρησιμοποιούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ως εγγύηση τα 10 δις που ούτως ή άλλως προβλέπονται για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Και επιπλέον, όπως θα ξέρετε με τον Επίτροπο Μπαρνιέ, ασχολούμαστε με την εξέλιξη του συστήματος για το κεφάλαιο κινδύνου. Και επίσης με το σχέδιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου προβλέπονται 2,5 δις ευρώ. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο στην συζήτηση με τα κράτη-μέλη θα το κάνει αυτό κατανοητό. Θέλουμε να αποδώσουμε αυτό το ποσό, αυτό το κονδύλι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης το εργαλείο αυτό του Venture Capital στις ΗΠΑ Πολιτείες έδωσε άριστα αποτελέσματα για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ στην Ευρώπη όχι ακόμη. Θα πρέπει να επιτρέψουμε αυτήν την εξέλιξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη, από τη σκοπιά της έρευνας και της καινοτομία με τον ορίζοντα το 2020. Για τον τουρισμό βρέθηκα την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, παρουσίασα την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ του τουρισμού και αύριο το πρωί στις 10 μέσω της γραπτής διαδικασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει ανακοίνωση που σκοπό έχει να χρησιμοποιήσει καλύτερα την ε, διαδικασία που ισχύει για τη χορήγηση θεωρήσεων και μετά την απόφαση του G20 που αφορούν τον τουρισμό ως εργαλείο κινητικότητας παγκοσμίω, εργαλείο καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη. Είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με το θέμα των θεωρήσεων, όχι μόνο από τη σκοπιά της ασφάλειας, αλλά ως αναγκαίο εργαλείο για την ανάπτυξη του τουρισμού και την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πρόταση που θα σημάνει την έναρξη σημαντικών αλλαγών σε αυτόν τον τομέα. Η πρόταση αυτή θα έχει την υπογραφή της Επιτρόπου Μάλστρομ και τη δική μου. Αύριο το πρωί θα λάβετε μόλις εγκριθεί το επόμενο δευτερόλεπτο το κείμενο της πρότασης. Διότι Επισήμω θα ακολουθήσουμε την κρατή διαδικασία και εφόσον όλοι οι βουλευτέ ε, που εργάζονται σε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και έχουμε και κάποιε επαφέ ε, μαζί. Ε, οπωσδήποτε θα λάβετε το κείμενο για την απελευθέρωση του χορήγηση των θεωρήσεων. Με την Επιτρόπο Δαμανάκη επίση συζητήσαμε προγράμματα τουρισμού για την Ελλάδα, ιδίω για τον τουρισμό στη θάλασσα, που αφορά ιδιαίτερο στην Ελλάδα. Οπότε από αυτή την άποψη θεωρώ ότι το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι χρήσιμο. Παρά την κρίση θα πρέπει να συνεχίσουμε. Ε, για την επαναφόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων η υπόθεση εξελίσσεται παράλληλα με αυτό που έθιξε η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, εγώ πάντοτε είμαι υπέρ της συμφωνίας μεταξύ των μερών. Όμως, αυτά τα μέρη δεν μπορούν λόγω κακής πίστης να αναβάλουν διαρκώς την λήψη απόφασης. Εάν κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν κάνει ένα βήμα πιστοχώρηση προκειμένου να προκύψει συμφωνία, εγώ δεν μπορώ να αποφύγω ε, να λάβω μια απόφαση που όμως δεν είναι στο δικό μου χέρι να την ε, αποφασίσω μόνος μου. Δεν μπορώ να αποφασίσω να ξεκινήσω έτσι μια νομοθετική διαδικασία. Αυτό αφορά και την επαναφόρτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και το ότι ισχύει για, τα, ε, για τον τομέα τη της γεωργίας και των τροφίμων. Σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα, η υπομονή μου έχει αρχίσει να εξαντλείται. Έτσι λοιπόν θα περάσουμε σε ένα impact assessment, σε μελέτη αντικτύπου και θα δούμε ποια θα είναι η απόκριση. Πρέπει να ξεκινήσει η νομοθετική διαδικασία με κάποιο τρόπο. Τώρα για το B2B, εκεί έχω ακόμη κάποια περιφόρια. Περιμένω να δω τι προτάσεις θα μου επιβληθούν. Η συνάντηση της 5 η ε, Δεκεμβρίου δεν θα είναι τελευταία, αλλά ελπίζω να προκύψει συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων, μεταξύ των μερών. Τώρα, αν και εσεί έχετε επαφέ με ε, του ενδιαφερομένους, πιέστε του να καταλήξουν σε ουσιαστική συμφωνία, γιατί πολλές φορές μιλάμε για συνένεση, συμφωνία και μετά επί της ουσίας αυτοί που λένε ότι υποστηρίζουν τη συμφωνία την υπονομεύουν και την υποσκάπτουν. Η, επί της αρχής θέση μου είναι η αρχής. Είμαι υπέρ της ε, ε, ε λήψης απόφασης και της, ε, του συστήματος της οικειοθελούς ε, συμφωνίας των μερών. Αλλά δεν μπορώ να είμαι σαν τον Πόντιο Πιλάτο και να ανύπτω τα σχήρας μου και να αφήνω να συζητιέται ότι βρέθηκε μια συμφωνία και τελικά μετά να μην υλοποιείται. Στον τομέα των, της γεωργίας και των τροφίμων είναι εξίσου σημαντικό το να βρεθεί μια συμφωνία όπως και για την ε, ηλεκτροδότηση. Θα δούμε λοιπόν τι θα αποφασίσουν και οι ενδιαφερόμενοι, οι μεν και οι δε. thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολλέ οι ερωτήσει που έπρεπε να απαντηθούν. Γι' αυτό θα παρακαλέσω του επόμενου συναδέλφου να συγκρατηθούν λίγο και να μην υποβάλουν πολλά ερωτήματα ταυτόχρονα. Στάιλερ, Κόζετσνικ, Σαλβίν, επόμενη. Θέλατε κι εσεί, κυρία Σαλντεμόζε. Το λέω. Ωραία. Και αυτή λοιπόν. Θα τη βάλουμε σε αυτό το γύρο. Ποια θα ξεκινήσει. Στάιλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Για τις οικοδομές είχα ένα θέμα. Είχατε έρθει πρόσφατα στη Σοσιαλιστική Ομάδα και μιλήσατε για τους ε, εμπλεκόμενους άρα θα συναντηθώ με εκπροσώπους του κατασκευαστικού κλάδου. Τι κάνει η Κομισιόν για να βοηθήσει την κατασκευαστική βιομηχανία, για να βοηθήσει την οικοδομή. Πραγματικά ανησυχούμε πάρα πολύ για το τι γίνεται στην πολύ σημαντική, στον πολύ σημαντικό αυτό κλάδο. Νομίζω δεν πέρασα τα 30 δευτερόλεπτα. Μπράβο σας, λέω πρώτος ο κύριος Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Φαντάζομαι ότι θα σας κάνουν δύσκολα ερωτήματα οι άλλοι συνάδελφοι. Εγώ έχω τρία ε, πολύ εύκολα σχόλια ε, για σας. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ για το ζήτημα της τυποποίηση, Είναι ένα πολύ σημαντικό για εμά θέμα και είστε ένα από αυτού που μας βοηθήσατε να θέσουμε το ζήτημα αυτό. Πριν από δύο χρόνια τώρα ξεκινήσαμε στο Στρασβούργο με κάποιους συναδέλφους κάποιες συναντήσεις. Και τώρα έχουμε μια πλατφόρμα, EU Growth Plan Dinner τη λέμε. Έχει μεγαλώσει η ομάδα μας, η παρέα μας και θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε και εσάς. Ο πρόεδρος συμμετέχει τακτικά στα γεύματα αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκλησή σας. Ε, για την αποδοχή της πρόσκλησης μάλλον και με ένα προσωπικό σχόλιο θα κλείσω. Είμαι υπεύθυνο για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και έχετε επισκεφθεί επανειλημμένως στη Λατινική Αμερική με αντιπροσωπεία επιχειρηματιών, εξ όσων γνωρίζω. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τι βλέπετε για το μέλλον των σχέσεων μας με τη Λατινική Αμερική. Ευχαριστώ. Σαλβίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Τρεις ερωτήσεις πολύ γρήγορες. Πρώτον, ετικετοθεσία και ετικέτες για τα εφαντουργικά. Δεν το συζητήσαμε στην ΙΜΚΟ γιατί μας είπαν ότι θα αναλάβει η Επιτροπή ΙΝΤΑ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε αυτό που έπρεπε, η Ολομέλεια αποφάνθηκε, αλλά μετά από δύο χρόνια σιωπής αποσύρθηκε η πρόταση. Δεν ξέρω λοιπόν το σακάκι που φοράω από ποια χώρα προέρχεται. Δεύτερη ερώτηση πώς σκοπεύετε να ασκήσετε πίεση. Διότι εγώ πιστεύω ότι ένας καταναλωτής έχει το δικαίωμα να γνωρίζει πού έχει παρασκευαστεί και έχει φτιαχτεί αυτό που φοράει και αυτό που αγοράζει. Επίσης για, τα, για τους διαγωνισμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες ενδιαφέρουσες προτάσεις αλλά προβλέπει στοιχεία αμοιβαιότητας για τις τρίτες χώρες και ιδίως για τις υπηρεσίες μέσω δημόσιων προμοθειών προμηθειών. Παρακαλώ διαβεβαιώστε με ότι δεν θα καταργηθούν οι ετικέτες ε, για τα ενδύματα, τα υφαντορκικά δηλαδή και για τα ενδύματα, διότι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, οι βαλτικές χώρες έχουν βάλει στο χρονοτούλαπο το θέμα αυτό. Επίσης για τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Η Ιταλία έχει αφαιρέσει, έχει εξαιρέσει τα δημόσια έργα από την νομοθεσία. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει να εξηγήσει μάλλον στα κράτη-μέλη ότι η εξαίρεση αυτή σημαίνει ένα σοβαρό ποσοστό καθυστερήσεων πληρωμών προς συγκεκριμένες τοπικές επιχειρήσεις. Πώς μπορούν να εξαιρούνται τα δημόσια έργα. Thank you very Ευχαριστώ πολύ κύριε και εσείς θα είσαστε πολύ γρήγορες φόλος. Πρόεδρε, ναι. Θα πρόκειται να μιλήσω σε ένα σεμινάριο για την ασφάλεια των προϊόντων σε μια ώρα. Ε, ρωτώ λοιπόν πότε σκοπεύετε να καταθέσετε αυτή την ε, δέσμη προτάσεων για την εποπτεία της αγοράς, κύριε Επίτροπε, στο Κοινοβούλιο, γιατί ασφαλώς οι παρευρισκόμενοι στο σεμινάριο θα ενδιαφέρονται. Επίσης για την ταξινόμηση των αυτοκινήτων, Πολύ καλά. Να μειωθεί η γραφειοκρατία όταν ε, μεταφέρουμε τι πινακίδε ενό. Παίρνουμε ένα αυτοκίνητο και αλλάζουμε πινακίδε από τον εκατό στο άλλο. Το θέμα όμω τη φορολογία. Σημειώνω δε ότι εγώ είμαι κατά τη αλλαγή του συστήματο φορολογία, γιατί είναι ζήτημα αρμοδιότητα των κρατών μελών, το αν θέλουν να φορολογούν τα αυτοκίνητα ή όχι. Αλλά πάντω πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία. Εγώ πρέπει να σας πω ότι αγόρασα ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στη Γερμανία, ε, Mercedes, και πρέπει να πω ότι το σύστημα στη, Γερμανία, στη Δανία για ταξινόμηση ήταν πολύ αποτελεσματικό. Πήγα 9 η ώρα το πρωί και μέχρι το 10 το μεσημέρι είχα νόμιμα μεταφέρει την, ε, το, τα χαρτιά του αυτοκινήτου στο σύστημα της Δανίας. Από ό,τι φαίνεται η γερμανική υπηρεσία λειτουργεί πολύ καλά. Ο κύριος ε, Στάμπ θα χαρεί. Εδώ λοιπόν το κείμενο που βάλαμε δεν προβλέπει φορολόγηση εναρμονισμένη. Όμω το κείμενο το εξετάζει αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο. Μπορεί λοιπόν να υποβληθούν τροπολογίε και να διορθωθεί αυτό. Το Κοινοβούλιο εδώ και 15 χρόνια είναι κυρίαρχο τη αποφάση και τη προτάσει αυτέ. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα τη ετικετοθεσία. Δεν αποσύρθηκε δεν αποσύρθηκε η πρόταση που αφορά τα ενδύματα, τα υφαντοργικά. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν ε, δύο εκθέσεις, μία για τις νέες απαιτήσει ε, της ετικετοθεσίας και έπειτα για τους ε, συσχετισμούς με τα αλλεργιογόνα, τι χημικέ ουσίε που μπορεί να χρησιμοποιούνται στα ενδύματα, κάτι που προβλέπεται και από την νομοθεσία περί φαντουργικών και ενδυμάτων που υιοθετήθηκε το 2011. Τώρα για το Made in το ζήτημα είναι λίγο πιο περίπλοκο. Όπω θα ξέρετε, ήμουν από του πρώτους υποστηρικτέ αυτή τη πρόταση από τότε που ήμουν βουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Και έπειτα, από το που συνέχισα και ανέλαβα κάθε κοντά επιτρόπου. Ο κύριος Αντεχουχτ ήδη είχε αποσύρει επισήμως την πρόταση, καθότι ο ΠΟΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, την είχε θεωρήσει ασύμβατη με τις εκεί διατάξεις. Ήταν ασύμβατη μετά του ΠΟΕ. Έπρεπε να σεβαστούμε και την απόφαση αυτή του ΠΟΕ. Άρα πρέπει να υποβληθούν νέες νομοθετικές προτάσεις με τρόπο εντός εισαγωγικών πιο ευφυή Δυστυχώς όμως, καθώς και η Ιταλία υπέβαλε μια νομοθετική πρόταση, όπου οριζόταν η προστασία του προϊόντος που κατασκευάζεται στην Ευρώπη ως απαράβατη αρχή, τελικά αυτό κόλλησε στο κοινοτικό επίπεδο. Για διαδικαστικούς λόγους ή για γραφειοκρατικούς κάποιες φορές θυσιάζεται μια τέτοια καθαγιασμένη αρχή. Πάντως η προάσπιση του Made in είναι πραγματικά καθοριστική σημασία για την προστασία και των προϊόντων μας και της παραγωγής της ε, ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Πάντως είμαι προθυμότατος να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε συνάντηση της ομάδας εργασίας του Κοινοβουλίου για την τυποποίηση Ας ορίσουμε μια ημερομηνία και με χαρά να ακούσω και τις δικές σας ιδέες και να δούμε τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε μαζί. Ακόμη και αν θέλουμε να ασχοληθούμε και με το πώ θα εξάγουμε τα δικά μα τα πρότυπα. Αυτό αφορά το δεύτερο μέρος, το σκέλος της ε, παρέμβασής σας. Ε, την Λατινική Αμερική ήδη είχαμε υπογράψει κάποιες συμφωνίες με χώρε της Λατινική Αμερική που έχουν να κάνουν με τα θέματα της τυποποίηση. Θεωρώ ότι η βιομηχανική πολιτική μα σε διεθνέ επίπεδο μπορεί να μα επιτρέψει να διερευνήσουμε νέες αγορές. Οι δικές μας επιχειρήσεις μπορούν αντί να μετατοπίζονται πλέον να, να λάβουν διεθνείς διαστάσεις, διεθνή δράση. Υπάρχουν σοβαρέ διμερεί συμφωνίε. Με τη Ρωσία είχαμε φτάσει στο 50%. Με τη Λατινική Αμερική επίση υπάρχουν δυνατότητε βιομηχανικών πρωτοβουλειών που μα επιτρέπουν να ε, δημιουργήσουμε καταστάσει για την παραγωγή ευρωπαϊκών προϊόντων για εκείνε τι αγορέ. Αυτό είναι σοβαρό. και μπορεί να τονώσει την πατρική ε, και μετρική επιχείρηση, για να το πούμε έτσι, δηλαδή την ευρωπαϊκή, με την Αργεντινή, τη Χιλή, την Βραζιλία, την Κολομβία, το Μεξικό, την Κεντρική Αμερική τώρα και τη Βόρεια Αμερική, αλλά τέλο πάντων κυρίως το Μεξικό, εκεί έχουμε αναλάβει δράση. Θα είμαι στο Περού στις αρχέ τη επόμενη χρονιά, οπότε σίγουρα θα τοποθετηθώ υπέρ των ε, συμφωνιών ε, τυποποίηση, των διμερών συμφωνιών τυποποίηση. Η Λατινική Αμερική είναι μια περίπτωση πολύ σοβαρή ε, για την ε, Ευρώπη. Εδώ και 15 χρόνια μας ε, απασχολεί αυτό το θέμα, διότι η Κίνα έχει αναλάβει δράση εδώ και κάνει πάρα πολλές επενδύσεις όπως συμβαίνει και στην Αφρική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν με τις προτάσεις για τη βιομηχανική πολιτική που εγκρίθηκαν πριν από τέσσερις εβδομάδες όντως θέλει να δώσει έμφαση στην διεθνοποίηση όπως έχει ονομαστεί προκειμένου να δοθεί μια νέα όθηση στην βιομηχανία μας. Σε ό,τι αφορά τη δεσμή μέτρων για την παρακολούθηση της αγοράς η πρόταση που είχε υποβληθεί εντός, θα έχει υποβληθεί έως το, εντός του 2013, το αργότερο το 2014. Με συγχωρείτε, λάθος. Μέσα στο 2012, το αργότερο αρχίζει το 2013. Ελπίζω λοιπόν μέσα στο φετινή χρονιά, το αργότερο την επόμενη, στις αρχές της επόμενης. Α, ναι, για τις δημόσιες προμήθειες, το ξέχασα δύο απαντήσεις εδώ για την αμοιβαιότητα και τις ε, βασικές αρχές. Νομίζω η απόκριση αυτή πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη. Κλασικά δίνω το παράδειγμα του ποδοσφαίρου. Επειδή είσαστε κι εσείς φύλαθλος. Δεν μπορεί να πηγαίνει κανείς στο Πεκίνο με ομάδα με λιγότερους παίκτες γιατί ούτως ή άλλως θα είναι σαν ένα το παιχνίδι. Όταν λοιπόν ο αντίπαλος έχει περισσότερες δυνάμεις πρέπει να είναι ανάλογος και αριθμό των παικτών, 9 προς 12 ας πούμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε ότι το νομοθετικό κείμενο της Ιταλίας μπορεί να μην συνάδει με τους κοινοτικού κανόνες, αλλά βεβαίω, εφόσον έχει εγκριθεί πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προσαρμοστεί το εθνικό νομοθέτημα. Α, ναι, και ο κατασκευαστικό τομέας. Για τον τομέα των κατασκευών, όπως θα γνωρίζετε, εγκρίναμε κείμενο πρόταση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οικολογικά συμβατές κατασκευές. Ο τομέας ο κατασκευαστικός έχει οριστεί ως τομέας προτεραιότητας για την βιομηχανική πολιτική. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτόν και να, απευθυνθούν εκεί και να κατευθυνθούν εκεί δημόσιες επενδύσεις, είτε κρατικές είτε ευρωπαϊκές. Έχει αποσταλεί επιστολή προς τα κατημέλη που τα καλεί να επενδύσουν και στην εξοικονόμηση, στην ε, ενέργεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα στην επάρκεια και εξοικονόμηση ενέργειας. Και τα project bond μπορεί να τονώσουν την, ε, τον κατασκευαστικό τομέα και τις σχετικές υποδομές με 17 δις ευρώ πρικοδοτήσαμε τον ε, τομέα αυτό προκειμένου να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές της ενεργειακής αποδοτικότητας και βεβαίως με την παρέμβαση της ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την ε, αποστολή κεφαλαίων και να μην αναγκαστούν τα κράτη-μέλη να να μην αναγκαστούν τα κράτη-μέλη να αποσύρουν τα φορολογικά κίνητρα που είχαν δώσει στον κατασκευαστικό τομέα τα προηγούμενα χρόνια. Παραμένει ένα τομέα προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά για να έχουμε μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ακούσουμε τους πέντε τελευταίους ομιλητές. Σύντομα παρακαλώ. Κορέα Δεκάμπος, Σφάπ, Βαλτασάρη, Μάιρ και η κυρία Ρούλα. Ναι, και εσάς, κυρία Ρίασα, ναι. Σας σημείωσα. Έξι. Άρα παρακαλώ, συντομότατα. Ξεκινάμε τον κύριο Αρίας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο που είναι σήμερα εδώ και για τη δουλειά που κάνει. Πολύ απαραίτητη και χρήσιμη. Σημαντικότατη ιδέα και για την κατάσταση που ζούμε σήμερα στην Ευρώπη και για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Για μια ακόμη φορά, Επίτροπε, θα ήθελα να σας μιλήσω για την ψηφιακή οικονομία. Πιστεύω ότι αναμφίβολα είναι ένα από τα ζητήματα για τα οποία πρέπει να ε, προωθήσουμε. Έχουμε ακούσει να λέγεται ότι είναι το μέλλον, είναι όμως και το παρόν. Πάνω απ' όλα λοιπόν και περισσότερο από ποτέ αυτή η βιομηχανική πολιτική πρέπει να διασυνδεθεί με τη νέα ψηφιακή εποχή, τις νέες τεχνολογίες. Και επομένω να είναι παρούσα η συνιστόσα αυτή στη νέα πολιτική. Μιλήσαμε για καινοτομία, εσωτερική αγορά. Αναφερθήκατε και στην ψηφιακή αγορά. Σας άκουσα επίσης να ε, μιλάτε για το Ολύμπιο. Φυσικά όλα αυτά περνούν από την νέα ψηφιακή εποχή, την νέα ψηφιακή τεχνολογία, το ίδιο και η περισσότερη Ευρώπη. Αν δεν έχουμε ψηφιακή διασύνδεση, δεν μπορούμε να έχουμε την περισσότερη Ευρώπη σε αυτό που θέλουμε. Απλούστευση. Το παράδειγμα που δώσατε με τις ταξινομήσεις ε, είναι πολύ επιτυχημένο. Δεν είναι όμως ε, αρκετό να απλουστεύσουμε τη γραφειοκρατία, που είναι σημαντικό βέβαια. Πρέπει όμως και να απλουστεύσουμε και να καινοτομήσουμε στο πλαίσιο της ε, νομοθεσίας. Γιατί τα πράγματα μας προσπερνούν, ε, πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από όσα θα θέλαμε και δεν έχουμε επιταχύνει στη νομοθεσία όσο θα θέλαμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε στους νέους καιρούς. Έχω μια υπόδειξη λοιπόν, όχι ερώτηση, σύνδεση με την ψηφιακή τεχνολογία. Αυτό θα μας βοηθήσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κύριε Σκορέντε, κάπως θα έχει το λόγο. Επίτροπε, είναι πάντοτε χαρά να σας έχουμε εδώ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι όλες ίσες. Ούτε ίδιες. Είναι πολύ διαφορετικές στον τρόπο που λειτουργούν, αλλά α πούμε ότι υπάρχουν δύο βασικέ κατηγορίε. Πρώτα απ' όλα οι συμβατικέ και κλασικέ που έχουν σοβαρά προβλήματα απασχόληση με του εργαζομένου και προβλήματα για τα οποία μπορούν να προβλεφθούν λύσεις, όπως είπατε με συγκεκριμένα προγράμματα όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά υπάρχουν και αυτές που είναι και Το εργαλείο αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να καλύψει και τις μεν και τις δε. Δεν μπορεί να είναι ίδια τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε για τις λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την έννοια της επιλογής ε, των διαφορετικών, λόγω των διαφορετικών κατηγοριών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ και τέσσερα χρόνια βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή, καμία παρέμβαση, εκτός από αυτή που ανακοινώθηκε, αλλά αυτό φαίνεται να είναι απλή προπαγάνδα και υποσχέσεις στον τομέα αυτό. Ως προς την ε, πραγματικότητα υπάρχει επιλεκτική πολιτική. Τι κονδύλια της Ευρώπης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των δύο κατηγοριών. Γιατί πραγματικά είναι σοβαρές οι διαφορές μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ κύριο Σφάπ. Ευχαριστώ πρόεδρε και σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο, κύριο Ταλιάνη, για τα όσα μας είπε, για τις προτάσεις ιδιαίτερα για τα τρακτέρ και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι χρειαζόμαστε τη δική του υποστήριξη για το Single Market Governance και τις προτάσεις του κύριου Μπαρνιέ όταν έρθει η ώρα. Χρειάζεται μια συνεργασία και για το σχεδιασμό αλλά και για την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και πάνω απ' όλα την υλοποίηση τις οδηγίες. Και ίσως χρειάζεται ε, μια ε, σύσταση αναχώρα για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτή. Περιμένουμε βέβαια την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαλτασάρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Προφανώς στηρίζω όλες τις πολιτικές που θα τονώσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την εθνοποίηση, την πρόσβαση στην επιστοπή, στις πιστώσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη λιγότερη γραφειοκρατία, την ανταγωνιστικότητα. Όμως θα βρισκόμαστε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Και έχω μια ερώτηση. Πώς μπορεί μια ε, μικρομεσαία επιχείρηση, με 30, 40, 50 εργαζομένους από την Ισπανία, την Ιταλία ή τη Γερμανία να ε, ανταγωνιστεί και να γίνει ανταγωνιστική στο επίπεδο της ε, ευρωπαϊκής αυτής αγοράς του μισού καταναλωτών. Είναι ωραίο όλο αυτό που λέμε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά λείπουν μεγάλες επιχειρήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως θα έπρεπε να υπάρξουν ανάλογες πολιτικές που να επιτρέπουν τη δημιουργία ομίλων, δικτύων, να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να οργανωθούν μεταξύ τους, ώστε να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό των διαστάσεων που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για να τονωθεί η ενία αγορά στην Ευρώπη, αλλά και για να κατακτήσουμε και νέες αγορές. Πώς μπορεί μια μικρή εταιρεία με 50 εργαζομένους να φτάσει στην Κίνα και στη Ρωσία ή ακόμα περισσότερο στη Βραζιλία και τη Λατινική Αμερική. Αυτές λοιπόν ε, οι μέρημνες μαζί με την ε, τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να μας δώσουν την προοπτική μιας εσωτερικής αγοράς πολύ πιο διευρυμένης και σε παγκόσμιο επίπεδο. Κύριε Σομπερμάια. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ. Καταρχάς, πρέπει να αξιολόγησες ότι ε, θα πρέπει να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από την καινοτομία. Και να αποφύγουμε τα κλεισίματα επιχειρήσεων όπως αυτή που ακούσαμε πρόσφατα για τη Γαλλία με 8.000 θέσεις εργασίας που θα χαθούν και άλλες 2.500 από την Όπερ. Ερωτούμε λοιπόν, τι μπορεί να γίνει ώστε να σταματήσει αυτή η φυγή. Η Αμερική, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, έχει κάνει πολλά για να διασώσει την αυτοκίνητο βιομηχανία της, αλλά παρενέβη και στις περιπτώσεις των μετατοπίσεων, μεταθέσεων παραγωγικών μονάδων. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχει κάποια ανάλυση, κάποιος κατάλογος, κάποιος άτλας, ώστε να καταγραφεί και τι σημαίνει χώρος παραγωγής, πώς ορίζεται δηλαδή και πώς ελέγχεται η διατήρηση του χώρου παραγωγής και επίσης γίνεται λόγος για εκατοντάδες χιλιάδες δισεκατομμυρίων περικοπές. Πώς είναι δυνατόν να κάνουμε περικοπές στα προγράμματα έρευνας όταν μιλάτε για δύο δις για την αυτοκίνητο βιομηχανία τα οποία θέλετε να διαθέσετε, δεν θα είναι τελικά αυτά χρήματα που θα στερηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ τελευταία και η κυρία Ρούλα. Ευχαριστώ. Δεν σχολιάζω τώρα τις προτάσεις. Περί αυτοκινητοβιομηχανίας και έτσι είναι υπερβολικά φιλόδοξα τα όσα μας είπε ο Επίτροπος. Λέμε δεν πας περιπτώσει, ένα πράγμα που ήθελα εγώ να αναφέρω, χωρίς να περιμένω απάντηση, ε, θέλω απλώς να το επισημάνω, το ζήτημα των κατεξουσιοδότηση πράξεων στον κανονισμό για τα ε, προϊόντα της κατασκευαστικής βιομηχανίας και οι προθεσμίες που προβλέπονται για την τήρησή τους. Έχουμε λοιπόν πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα αυτών, οι οποίες μου έχουν ε, επισημάνει πως υπάρχουν πολλά προβλήματα από τις καταξιδότητες πράξεις που περιμένουν να λειτουργήσουν, να δαθούν σε εφαρμογή και επίσης πολύ φοβούμαι ότι θα ξαναρχίσει η συζήτηση που είχαμε και με τα παιχνίδια στα βαρέα μέταλλα ή στις, ε, στην ηχορύπανση θα έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, καλό θα ήταν μια και έρχονται Χριστούγεννα και ασφαλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ενημερωθούν, θα ανακοινήσουν το θέμα αυτό της ασφάλειας των παιχνιδιών, καλό θα ήταν να μην το παραλείψουμε. Ο Επίτροπος, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σας, όσο μπορείτε παρακαλώ θα μας διαθέσετε με τις απαντήσεις σας. Θα χρειαζόταν ένα μισάωρο για να παρουσιάσω λεπτομερώς και καταλεπτός την πολιτική που θέλουμε να καταρτήσουμε για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ιδίως τις στιγμές αυτές της κρίσης είναι πολλές οι μεγάλες εταιρείες αλλά και χιλιάδες οι μικρότερες που υποφέρουν λόγω της κρίσης στην αυτοκινητοβιομηχανία. Την Παρασκευή το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ένα τελικό κείμενο της ΚΑΡΣ 21 και θα είναι και ένα σχέδιο δράσης για το αυτοκίνητο για τα ερχόμενα χρόνια. Θα επικεντρωθούμε σε τρεις βασικές πτυχές. Πρώτα απ' όλα την ευφυή ρύθμιση ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις σε αυτές τις σημερινές συγκυρίες να αντέξουν την υπέρμετρη πίεση σε όλους τους τομείς. Βεβαίως δεν θα απαρνηθούμε τις προσπάθειές μας για την αναχέτηση των κλιματικών αλλαγών, για τη ρήπανση, όμως θα δείτε ότι το κείμενο που θα εγκριθεί την πέμπτη το πρωί θα πετυχαίνει μια σωστή ισορροπία μεταξύ της περιβαλλοντικής πολιτικής και της βιομηχανικής μας πολιτικής, ακόμη και σε ό,τι αφορά τις ρυθμιστικές στοιχές, σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση. Θα προτείνω στο ερχόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να περάσουμε από το σημερινό δις επενδύσεων για την κοινοτομία και έρευνα στον τομέα του αυτοκινήτου, της αυτοκινητοβιομηχανίας, στα δύο δις, 15 δύο δις για το πράσινο, το οικολογικό δηλαδή αυτοκίνητο του μέλλοντος, για να υπάρξουν εδώ και απαραίτητες επενδύσεις στην κοινοτομία και έρευνα. Οι παρεμβάσεις που θα δίνουν κίνητρα, όχι ο κρατικός προστατευτισμός, η παροχή κινήτρων προς τους πολίτες για την αγορά αυτοκινήτων που δεν ρηπαίνουν, είναι κάτι που προφανώς δεν θα μας βρει αντίθετος. Επίσης, για την εμπορική μας πολιτική. Εδώ μπορούμε να είμαστε αφελείς. Γι' αυτό αποφασίσαμε να έχουμε και κάποιες αποφάσεις περί ανταγωνιστικότητας πριν την υπογραφή των διεθνών μας συμφωνιών. Ξεκίνησε μάλιστα μια μελέτη για τις διεθνείς ε, συμφωνίες που έχουμε προσυπογράψει για να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπό τους και όπως θα γνωρίζετε η βιομηχανική μας πολιτική και η εμπορική πολιτική προβλέπει την ε, η λειτουργία παράλληλων ε, task force, ομάδων ε, δράσης για τη βιομηχανία και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, ώστε ετησίως να εντοπίζεται η πολιτική δράση που πρέπει να υλοποιηθεί για την ε, βιομηχανία μας. Εδώ θα ασχοληθούμε και πάλι κατά προτεραιότητα με τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Επίσης, έλαβα επιστολή από 7 υπουργού των ε, μηχανικών υποθέσεων των κρατών μελών ε, και μου ζήτησαν να συναντηθούμε για να συζητήσουμε για την κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη πριν από το επόμενο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. Εκεί θα συζητηθεί και το ΚΑΡΣ 21, αλλά θα ξεκινήσει συζήτηση και για την κατάσταση της αυτοκινητοβιομηχανίας καθώς και το σκέλος της ανταγωνιστικότητάς της στην Ευρώπη. Επιπλέον, ήδη αποφάσισα πριν τα τέλη Νοεμβρίου να συναντηθώ με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και των Ευρωπαϊκών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για να δούμε ακριβώς αυτό το ζήτημα. Θα ακούσω λοιπόν πέρα από τις στατικές δράσεις που θα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα δράσης που θα εγκρίνει το Κολέγιο των Επιτρόπων μεθαύριο, πέραν αυτού θα μελετήσουμε το τι μπορεί να γίνει βραχυπρόθεσμα. Δεν πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να παρέμβει στι αρμοδιότητε των κρατών ούτε το τι καθορίζουν για τι μεμονωμένε επιχειρήσει. Όμω, ενώπιον μια τόσο οξία κρίση που πλήττει τον τομέα τη αυτοκινητοβιομηχανία, θα πρέπει να μπορεί να αναλάβει πλήρω το ρόλο τη ω συντονίστρια. Συντονίστρια των πολιτικών, διότι το σύστημα, ακριβώ όπω έχει ζητηθεί και από τη βιομηχανία, και από τα κράτη-μέλη, αυτό ακριβώς θα πρέπει να μπορεί να φέρει πέρα έναν ενεργό ρόλο. Δεν θέλουμε να παραβιάσουμε τους κανόνες, ούτε να παρέμβουμε στην ε, ελευθερία των κατών μελών, όμως θέλουμε να υπάρξει έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να υπάρξει ένας βιομηχανικός γάμος της ε, βιομηχανίας και του αυτοκινήτου. Καθοριστική σημασία για να ξεφύγουμε από την κρίση είναι από τους πρώτους τομείς που έχουμε ορίσει ως ε, τομέα προτεραιότητα στη νέα μα βιομηχανική πολιτική. Βιομηχανική πολιτική η οποία θα πρέπει να περάσει και σε έναν εξυγχρονισμό με την ανοτεχνολογία, λόγω χάρη, με την ε, ψηφιακή διάσταση, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το e-commerce, τις συναλλαγές με ηλεκτρονική υπογραφή. Όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τον εξυγχρονισμό τρίτη βιομηχανική επανάσταση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ψηφιακή οικονομία στο κέντρο της. Θα συμφωνήσω λοιπόν εδώ με τον κύριο Σφάμπ. Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλήθεια είναι ότι σήμερα μόνο το 13% μπορούν να δραστηριοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μικρό ποσοστό επίσης εκτός της χώρας προέλευσής τους. Κάνουμε προσπάθειες και προς αυτή την κατεύθυνση και σκέφτομαι εδώ τις ε, επανειλημμένες προσπάθειες των κλάστες, επίσης των δημοσιονομικών ε, εργαλείων που αφορούν την κατάρτιση και εδώ χρειάζεται μια ευρύτερη στρατηγική ούτως ή άλλως. Τα δίκτυα των επιχειρήσεων. Εδώ στην Ιταλία το ανάλογο πρότυπο λόγω χάρη μπορεί να φαίνεται ήδη κάπως ξεπερασμένο αλλά για την διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπάρχει έγγραφο που αφορά ακριβώς την εξωτερική λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχει εγκριθεί εδώ και κάτι μήνες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς η τόσο μεγάλη επικοινομορφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ανάγκη να αναπτυχθούν και να συνεργαστούν μεταξύ τους για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες βιομηχανίες, όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τη ε, διαφοροποίηση της χρηματοδότησης. Αυτό δεν, ε, που θυμήσατε δεν ήταν μόνο προπαγανδιστική κίνηση. Τα 13 δις ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2009 εντάξει ήταν ένα θέμα. Όμως στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα είναι σαφές το τμήμα το σκέλος καινοτομία έρευνα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει εντό του ορίζοντα 2020 και το τμήμα ανταγωνιστικότητας και τουρισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο ε, πακέτο δέσμη, ε, κόσμε, συγγνώμη, εντός ε, που θα είναι περίπου στα 2,5 δις ευρώ. Για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, για τα γεωργικά προϊόντα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις αλλά για τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να σας ενημερώσω γραπτός ε, εντό των επόμενων ημερών, προκειμένου να ξέρετε και το ακριβές πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι απ' έξω. Η ηλικία μου επιβάλλει και κάποιους τέτοιους περιορισμούς. Δυστυχώς προχωρά αυτή. Νομίζω ότι απέντησα σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις. Θα είμαι στη διάθεσή σας ακόμη και για κατηδίαν συναντήσεις. Και ελπίζω στη συνεργασία της Επιτροπής σας και για την βιομηχανική μας πολιτική και για την εσωτερική αγορά γενικότερα. Θυμίζω ότι αύριο θα εγκριθεί από το Κολέγιο των Επιτρόπων η ανακοίνωση για τις θεωρήσεις, κάτι πιστεύω ιδιαίτερα χρήσιμο και σημαντικό για την κυκλοφορία των ε, πολιτών εντός της αγοράς και μεθαύριο το πρόγραμμα δράσης για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ολοκληρώνεται το έργο της ΚΑΡΣ 21 και τις επιμέρους λεπτομέρειες για τις πρωτοβουλίες μετά τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των κυβερνήσεων θα τα ανακοινώσω, θα τα δούμε μαζί και θα τα συζητήσουμε ώστε να καθορίσουμε την ε, πορεία μας και να δούμε τη διάσταση όχι μόνο της βιομηχανίας αλλά της κοινωνικής πολιτικής οι συνάδελφοι Αλμούνια και Άντερ θα ε, συνεργαστούν μαζί μου ώστε να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική, πολιτική εσωτερική αγορά, αλλά ταυτόχρονα και κοινωνική. Έτσι θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε την Ευρώπη από την κρίση με τέτοια στρατηγική σημασία μέσα. Επίτροπε Ταγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ που απαντήσετε τόσο καλά σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Σας αξίζει ένα ζεστό χειροκρότημα. And, um, I Και νομίζω ότι το επίπεδο των ερωτήσεων δείχνει πόσο μας ενδιαφέρει ιδίω ε, η βιομηχανική πολιτική ορισμένη τομή τη και θα συζητήσουμε και με του συντονιστέ αργότερα πώ μπορούμε να δώσουμε πιο θαραλέα απάντηση, να βρούμε απαντήσει στην Επιτροπή μα, αλλά και βέβαια και η Επιτροπή Βιομηχανική Πολιτική. Θα περιμένουμε λοιπόν τις μελλοντικές ανακοινώσεις σας. Ε, ήταν μεγάλη χαρά που σας είχαμε εδώ και προσβλέπουμε στην επόμενη επίσκεψή σας. Now for the next item, um... Για το επόμενο ζήτημα θα προεδρεύσει η κυρία Βερνιώτη, πρόεδρος. Και θα επανέλθω εγώ στις 5 για τη συνεδρία των συντονιστών. Λοιπόν, πριν μιλήσαμε για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τώρα θα εξετάσουμε την έκθεση του κυρίου Χατζημαρκάκη. Γνωμοδότηση λοιπόν ακριβώς για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή και μετά στους κοιόδης εφόσον παρίστανται. Δεν βλέπω και πολλού μέχρι στιγμή στην αίθουσα, αλλά τέλο πάντων. Όλοι εδώ είναι, μπράβο. Τέλο πάντων και όσοι έρθουν ευπρόσδεκτοι. 20-25 λεπτά άντε έχουμε. Λοιπόν, κύριε για αυτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κατέστησε σαφέ ο Επιτροπό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά προγράμματα δράσεω. Το πρόβλημα μα είναι ότι δεν είναι ορατά στον πολίτη. Και το πρόβλημα είναι εν τέλει ακριβώς αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται ο πολίτης. Αυτό έχει σημασία. Συζητήσαμε ήδη και για την ανάγκη και δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας στην νέα αγορά. Βλέπουμε δυστυχώς ότι μπορεί κάποιοι να πιστεύουν σε αυτή την προοπτική, αλλά ιδιαίτερα στις χώρες που πλήττονται βαρύτατα από την ε, ανεργία, η δυσπιστία είναι πολύ μεγάλη. Και έτσι χρειάζεται να στηριχθούμε και να αναπτύξουμε την ιδέα της πρόσβασης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω των εθνικών τραπεζών επενδύσεων, οι οποίες θα πρέπει και να δημιουργηθούν αν δεν υπάρχουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η KFA γερμανική, η πιστοτική το, το, Ίδρυμα για την Ανασυγκρότηση είχε θεσπιστεί την εποχή του σχεδίου Μάρσαλ με κονδύλια του σχεδίου Μάρσαλ και μπόρεσε να βοηθήσει ε, για την πρόοδο και την ανασυγκρότηση στη Γερμανία. Εάν το είχαμε αυτό σε θέση μας, θα μπορούσαμε να είχαμε βοηθήσει σημαντικά κράτη όπως η Ουγγαρία ή η Ελλάδα. Δεν θα είχαν πληγεί τόσο βαριά από την κρίση του. Μεταξύ έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν έχουμε μπορέσει να προχωρήσουμε σε ουσιαστική στήριξη. Γι' αυτό λοιπόν και προτείνω με τις ε, τροπολογίες τις οποίες έχω δει και για τις οποίες ευχαριστώ συναδέλφους ε, τα εξή. Υπάρχουν ε, τροπολογίες για την παράγραφο 2 του κειμένου μου όπου κυρίως σαν τροποποίηση προσφέρεται η, συμπλήρωση του κειμένου με νούμερα, με αριθμητικά στοιχεία για τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις που καθίσουν πιο ορατά και πιο κατανοητά αυτά που θέλουμε να πούμε. Για την παράγραφο 3 υπάρχουν πολλέ τροπολογίε, ιδιαίτερα για το συσχετισμό μεταξύ τραπεζών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις σχέσεις μεταξύ τραπεζών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορούν να διαδραματεύσουν, να διαδραματίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λόγω της ε, ποικιλία στις Ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα τις εξετάσουμε. Στο, στην παράγραφο 5 κυρίως ε, έχουμε να κάνουμε τις Εθνικές Τράπεζες Επενδύσεων και πάλι έχουμε τροπολογίες εδώ από δύο κυρίως συναδέλφους και από τον πρόεδρο που ιδιαίτερα υπογραμμίζουν το θέμα των λεγόμενων business angels, ένα μέσο χρηματοδότησης όχι καινούριο, αλλά πολύ καινοτόμο για ορισμένες χώρες, και που μπορεί να διδερματίσει ιδιαίτερα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Χαίρομαι ιδιαίτερω για τι τροπολογίε που είδα εδώ. Παράγραφο 6. Γίνεται λόγο για καλύτερη, για πιο πλήρε και έγκυρε πληροφορίε. Χαίρομαι ιδιαίτερω. Πολλοί συνάδελφοι θέλουν να διευκρινίσουν το κομμάτι αυτό και προτείνουν μια ενιαία ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσε να αποβεί εις όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί είναι πολλές οι δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξει. Επίσης, μέσα χρηματοδότησης και κατάρτιση είναι αντικείμενο τροπολογιών που δεν ξέρω αν είναι θέμα δικής μας αρμοδιότητας, αλλά εν πάση περιπτώσει συμφωνώ με τις ιδέες. Παράγραφος 7. Γραφειοκρατικό άχθος. Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα επιβαρύνονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις από αυτό. Αν χρειάζεται, παραδείγματι, να δαπανίσουν πολύ χρόνο για μια ε, διατύπωση γραφειοκρατική. Άρα λοιπόν ε, μείωση της γραφειοκρατίας, ιδιαίτερη υποστήριξη στις ε, μικρομεσαίες που ξεκινούν και το καθεξής. Παράγραφος 8, καθυστέρηση πληρωμών, θέματα που συζητήσαμε τώρα και με τον Επίτροπο. Με ικανοποίηση σημειώνω ότι μας ε, προσχέθηκε την υποστήριξή του. Έχουμε επίση μια τροπολογία για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ιδιαίτερως για την ε, κατάρτιση αξιόπιστων επιχειρησιακών σχεδίων, business plan. Συμφωνώ και στην 10 που γίνεται λόγος για ε, δίκαιο και διαφορά σε νοσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο και πρόσβαση. Ίσως να γνωρίζουν κάποιοι συνάδελφοι ότι έχει το ελεγκτικό συνέδριο καταθέσει έκθεση πρόσφατα για τις αθέμητες πρακτικές ορισμένων κρατών ως προς το ε, ρυθμιστικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να μην γίνεται πιο οικονομική αξιοποίηση των πόρων χωρίς αυτή να είναι παράνομη απαραίτητα. Γι' αυτό λοιπόν στις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να μεριμνήσουμε αυτήν την δική μας δουλειά ώστε να γίνονται σωστά οι αναθέσεις ε, και βέβαια να υποφελούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υπάρχει εποπτεία, όλα αυτά που έχουν με στη συζήτηση και με τις δημόσιες προμήθειες. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους που κατάθεσαν τροπολογίες και είμαι στη θέση για τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε κύριε Χατζημαρκάκη. Οι σκιώδες λοιπόν έχουν το λόγο για το ΕΛΚ η Μαργαρίτα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας. Να τον ευχαριστήσω θερμά για το έργο του. Συμφωνώ με τις γενικές κατευθύνσεις στο γενικό προσανατολισμό που μας παρουσιάζει και συμφωνώ με όσα είπε. Πιστεύω ότι θα πρέπει ειδικότερα να τονίσουμε την απλούστευση της πρόσβασης ε, στις πληροφορίες, ένα ζήτημα που ανέφερε ο συγκητή. Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ενημέρωση, δηλαδή για τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει έλλειψη πληροφοριών που πολύ συχνά αποτελεί φραγμό που δεν επιτρέπει τη σωστή χρήση της χρηματοδότησης. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε εκ νέου ε, την εμπιστοσύνη προς τους ε, δανειδοτικούς οργανισμούς που δεν είναι τόσο πρόθυμοι να δώσουν πια χρηματοδότηση. Υπάρχει όμως ένας ολόκληρος κλάδος μικρομεσαίων επιχειρήσεων που λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης απελπίζονται και δεν επιδιώκουν αυτή τη χρηματοδότηση. Υπάρχει έλλειψη λοιπόν εμπιστοσύνης προς τους δανειοδοτικούς οργανισμούς και αυτό είναι σημαντικό. Να επισημάνω και ένα ακόμη θέμα. Ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσει θα πρέπει, οι, συγγνώμη, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα πρέπει να γίνουν πιο επαγγελματικές δηλαδή στην προσέγγιση τους, θα δημιουργήσουν επιχειρησιακά σχέδια να βελτιώσουν ε, τις δυνατότητέ τους. Οι επενδύσεις θα αυξηθούν αν οι επενδυτές που πολύ συχνά έλκονται από τα κέρδη, αν πιστούν λοιπόν οι επενδυτέ αυτέ ότι μια δεδομένη εταιρεία μπορεί να αναπτυχθεί, ότι έχει δυναμικό, αναπτυξιακό δυναμικό και μπορεί να παραγάγει κέρδο, θα είναι θετικό. Και πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν την ελκυστικότητα των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς τους ε, επενδυτές. Πολύ σημαντικός επίσης είναι ο ρόλος που έχουν τα πιστικά επιχειρηματικά σχέδια από πλευράς ΜΜΕ. Διασφαλικές επενδύσεις. Υπάρχουν εμπόδια. Πρέπει να τα καταρρύψουμε, συμφωνώ με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπάρχει ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο και δι φορολογία. Η διπλή φορολογία, για παράδειγμα, που τρομάζει τις ΜΜΕ και τις αποτρέπει από το να προσπαθήσουν να διεισδύσουν στην αγορά άλλων χωρών. Έχουμε μια σειρά τροπολογιών και σε σχέση με το ΦΠΑ και την απλούστευση του συστήματος αυτού που είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα επίσης. Όχι το μόνο όμως. Δεν είναι το μόνο θέμα που εκκρεμεί. να το αναφέρουμε μεν μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο, αλλά όχι ως το μόνο ζήτημα που είναι ακόμη σε κρεμότητα και πρέπει να επιληθεί, να αντιμετωπιστεί για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Συνοψίζοντας, ευχαριστώ για ακόμη μια φορά τον εισηγητή για την πολύ καλή του δουλειά και πιστεύω ότι θα είναι πολύ αποδοτικό ζήτημα που θα το χειριστούμε με πολύ καλό τρόπο, πολύ θετικό και έτσι αυτό θα αποβεί προς όφελο και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ την κυρία Χάντσλικ. Ο Αντώνιο Φερνάντο Κορέα Ντεκάμπος έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες είναι όντως η ναυαρχίδα της παραγωγικής μας βιομηχανίας. Με 80% των θέσεων εργασία. Πρέπει λοιπόν να τις κοιτάξουμε προσεκτικά. Κάθε μία από αυτές έχει διαφορετικά, διαφορετικές δυνατότητες και συμφέροντα. Υπάρχουν κάποιες παραδοσιακές, θα λέγαμε, οι οποίες παρακολουθούν τις παραδοσιακές μεθόδους εργασιακές και παραγωγικές και άλλες καινοτόμε που εκτίθενται διαφορετικά στον ανταγωνισμό. Οι δυνατότητες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα κράτη-μέλη στην δημοσιονομική ανασυγκρότηση μπορεί να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις και κυρίως για τις θέσεις εργασία, αλλά και για τον καταναλωτή. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα μία σειρά μέτρων με δυνατότητα πρόσβαση σε, ευρωπαϊκή, σε εθνική αλλά και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και θα έπρεπε να γίνει μία μελέτη συνεπειών των μέτρων αναδιάταξης των δημοσιονομικών στα κράτη-μέλη ώστε να αξιοποιηθούν νέε ευκαιρίε για χρηματοδότηση, κυρίω μέσω των business angels, όπω υπόθηκε νωρίτερα, και να κοιτάξουμε τι νέε πρακτικέ, τι βέλτιστε πρακτικέ για την μείωση της ε, γραφειοκρατίας πάνω απ' όλα. η δική μου ιδιαίτερη η πατρίδα έχει μια πολύ καλή επίδοση. Μπορεί μέσα σε 23 λεπτά, λιγότερο από μισή ώρα, να δημιουργήσει κανεί μια μικρομεσαία επιχείρηση. Αυτό θα πρέπει να είναι ο μέσο όρο στην εσωτερική αγορά. Με εντυπωσιακό, κύριε Κορέιρα κάπω, Αλλά άπαξ και ιδρύθηκε η επιχείρηση, τι γίνεται. Κυρία Ρούλε, αν δεν με, έχει στήσει το λόγο εκ μέρου του Πρασίνου. Πρόεδρε, εμείς δεν έχουμε τροπολογίες ε, διατυπώσει. Εγώ δηλαδή, γιατί έχω τόσο πολλή δουλειά με άλλες εκθέσεις που δεν πρόλαβα. Είναι πολύ καλή η εκθέση σας κύριε Χατζημαρκάκη. Θέλω απλώς να επισημάνω ότι υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που επίσης θεωρώ εξαιρετικές επί παραδείγματι την υπαριθμών 12, η οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει περισσότερη συνέπεια μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων που ε, υποβάλλει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι ξαφνικά όλοι οι επίτροποι ανακαλύπτουν τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, πράγμα το οποίο βέβαια δυσκολεύει την ε, επισκόπηση όλη τη κατάσταση. Δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση. Κάθε ένας προσπαθεί να βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά από τη δική του πλευρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, με τις Εθνικές Τράπεζες Αναπτύξεως Ίσως θα έπρεπε και να αναφέρουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία δεν αναφέρεται στο κείμενο. Με όλες τις πεκκίσεις που μπορεί κανείς να έχει, είναι μια τράπεζα ευρωπαϊκή, η οποία στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως μικρά ε, έργα, μικρά σχέδια. Ίσως λοιπόν συμβαστικά ενδεχομένω να μπορούσε να ενσωματωθεί. Πάντως εν γέννη είναι καλή έκθεση. Και ο κύριος Μπίλαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους της κυρίας Μακλάρκιν, η οποία λόγω άλλων σημαντικών δεσμεύσεων στην εκλογική της περιφέρεια δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή για την έκθεσή του, είναι πολύ καλή. Η κυρία Μακλάρκιν έχει καταθέσει κάποιε τροπολογίε για να ενισχύσει το κείμενο περαιτέρω. Έχει υπογραμμίσει η κυρία Μακλάρκιν τη σημασία τη ε, βελτίωση τη ενημέρωση και τη πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τι πηγέ χρηματοδότηση. Έχει υπογραμμίσει τη σημασία των ε, κρατών μελών και του ρόλου τους στο να στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε να και τις λάβουν υπόψη σε κάθε τομέα πολιτικής. Επίσης υπάρχει μία ε, τροπολογία για ένα σύστημα εποπτείας ώστε να εξασφαλίζεται ότι θα ε, λειτουργεί το σύστημα πρόσκοπτα στην ε, δανειοδότηση των τραπεζών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι οι συνάδελφοι έλαβαν το λόγο. Ας ακούσουμε τον κύριο Χατζημαρκάκη. Πρόεδρε, ευχαριστώ για το φόρο προσθέμενης αξίας της κυρίας Χάντσλικ. Θα ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχει μια καλή τροπολογία της κυρίας Μακλάρκιν ή παρελθμόν 28 την οποία και εγώ συμμερίζομαι, γιατί συμφωνώ μαζί το πρόβλημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι ο φόρος προσθέμενης αξίας μόνο. Είναι πολλά άλλα τα προβλήματα, αλλά είναι κατά κύριο λόγο φόρος προσθέμενης αξίας. Άρα λοιπόν κάποιες ιδέες της κυρίας Μακλάρκιν τις δέχομαι και τις ενσωματώνω. Πάντως, όπως είπα, με ελάχιστε εξαιρέσει, είναι πάρα πολύ καλές οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και θα της ενσωματώσουμε στο κείμενο στο βαθμό που γίνεται. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάρχουν δυνατότητες όντως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δραστηριοποίηση με μέσα που γνωρίζουμε από το Just Πασφερρυπίνη, το Jeremy, το Risk, share, risk Shared Finance Facility, άλλα μέσα δηλαδή χρηματοδότησης, γιατί διαχειρίζεται κονδύλια από του τομεί Φερρυπίν τη έρευνα ή τη περιφερειακή ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων και με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζει πρόσβαση για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ή διευκολύνει την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τέτοια χρηματοδότηση. Γι' αυτό και έχει αποδείξει, όπως έχω επισημάνει, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ότι λειτουργεί το σύστημα αυτό. Θα δεχθώ την προσβαση των μικρομεσαιων επιχειρησεων σε τετοια χρηματοδοτηση γι αυτο και εχει αποδειξει όπω εχω επισημανει η ευρωπαικη τραπεζα επενδυσεων οτι λειτουργει το συστημα αυτο θα δεχθω την προταση και θα το ενσωματώσουμε. αλλά πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιληφθεί η ίδια ότι συμβαίνει αυτό. Γιατί κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Είναι πολλά τα ποσά και μεγάλα τα ποσά. Φερρυπίν, πρόγραμμα για την Ελλάδα. 10 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία βρίσκονται στους ε, λογαριασμούς και κοιμούνται χωρίς να απορροφούνται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκατοντάδε φορέ έχει πει ότι υπάρχουν, αλλά φαίνεται ότι στι Βρυξέλλε οι γραφειοκράτε, όχι στο Λουξεμβούργο που είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά στι Βρυξέλλε φαίνεται ότι κοιμούνται βαθιά οι υπάλληλοι τη Επιτροπή. Ε, βλέπω λοιπόν με πόνο καρδιά να ε, υποφέρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά του, που κλέβουν οι επιχειρήσει του, γιατί δεν διατίθεται κονδύλια εφιστάμενα. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι όλοι σημειώσατε το επαντλημένο αίτημα, το επίμονο αίτημα και σίγουρα η διακρατική συνεργασία αλλά και η συνεργασία κρατών και κοινοβουλίου και κομισιών είναι κάτι που πρέπει να γίνει και εμεί πρέπει να πιέσουμε, πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα για να προχωρήσουμε λίγο ταχύτερα. Έχουμε μείνει πολύ πίσω και καιρό είναι να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι στην καρδιά της ανάπτυξης. Δεν μπορούμε να περιμώσουμε ε, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Μόλις πέντε και κυρίως ο τη συνεδρίασης. Ε, πέντε και κλεισμένα των θερών συνεδρίαση των συντονιστών. Ευχαριστώ.